αύριο ε, στις 12 το μεσημέρι. Η ημερήσια διάταξη μας οδηγεί τώρα στην κοινή συζήτηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να ξεκινήσω θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά την κυρία Μακέντάιρ. Thank you, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συζήτε για το ιδιαίτερα επικοδομητικό έργο του σε σχέση με την έκθεσή μου. Επίσης χαιρετίζω την σημερινή κοινή συζήτηση ε, μαζί με την πρωτοβουλία ε, για, τα 10, για τις 10 ενέργειες από την Επιτροπή Ήτρε που συμπληρώνει τη δική μου έκθεση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για να αντιμετωπίσουμε τα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσουμε νέους καινοτόμους τρόπους κατά τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει δημιουργία ενό περιβάλλοντο υποστηρικτικού προ τι επιχειρήσει που θα δίνει εμπιστοσύνη στι επιχειρήσει αυτέ ώστε να επενδύουν και να μεγαλώνουν. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι ει βάρο τη ε, υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση αυτή. Δική μου φιλοδοξία δεν είναι να μειώσουμε το επίπεδο προστασία των εργαζομένων ή τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά να μειώσουμε τη γραφειοκρατία διευκολύνοντας την κατανόηση και την υλοποίηση της νομοθεσίας, βελτιώνουμε τη συμμόρφωση και την ασφάλεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε το σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα προστατεύει τους εργαζομένους και ταυτόχρονα θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξάνονται, να καινοτομούν και τελικά να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε δει ότι έχει γίνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση με την πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιο πρόσφατα για το τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την πρωτοβουλία των 10 μέτρων που έχει εντοπίσει τις 10, τα 10 νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβαρύνουν περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ευρύτατο το πλαίσιο των θεμάτων που μας απασχολούν στην έκθεση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι τελικά καταλήξαμε σε μια σωστή ισορροπία. Έχουμε συμφωνήσει σε πολλά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα και την καλύτερη νομοθεσία η βάση αυτής της έκθεσης είναι το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, αυτή τη στιγμή παρέχουν 90 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ε, στον ε, ιδιωτικό τομέα και υπάρχει μια οργάνωση που εκφράζεται υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που είναι η, κυρί, η κύρια οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και καλούν τους Ευρωπαίους πολιτικούς ε, εν ώψη των εκλογών που επίκυνται ε, και λένε ότι η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στην καρδιά της ανταγωνιστικής Ευρώπης σε ένα κόσμο ταχαίως αναπτυσσόμενων οικονομιών το να δημιουργεί κανείς δική του επιχείρηση είναι κάτι που δίνει έμπνευση και συνεισφέρει προς την, στο οικονομικό περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας για να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις ε, και να επιβιώσουν και να αυξάνονται και να είναι ανταγωνιστικές μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αυτό σημαίνει επένδυση σε δεξιότητες, σημαίνει ευέλικτη νομοθεσία που θα είναι διαχειρίσιμη και θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, δίκαιο πεδίο ε, ε, για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν 90 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και απασχολούν τα 2 τρίτα των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταρχήν στις πολιτικές για την απασχόληση. Στην έκθεσή μου λοιπόν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα είναι ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καλύπτει διάφορους τομείς. Το κόστος και η πολυπλοκότητα της έναρξης μιας επιχείρησης πρέπει να μειωθούν. Οι δεξιότητες είναι σημαντικές για, για το εργατικό δυναμικό που θα πρέπει να είναι δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται η αγορά, επιχειρηματικότητα οι νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση από 45% έχουν μειωθεί στο 30% τα τελευταία τρία χρόνια. Θα πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία του παρελθόντος και η έκθεσή μου καλύπτει και δημογραφικά στοιχεία και θέματα πρόσβαση στην αγορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καλύτερη νομοθεσία. Όλα αυτά τα θέματα καλύπτονται στην έκθεσή μας. Μαζί με άλλους 84 ευρωβουλευτές Υποβάλλουμε μια τροπολογία για την Ολομέλεια, την οποία ελπίζω ότι μπορείτε να υποστηρίξετε. Η τροπολογία υπαριθμών 2 τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ε, πολλές θέσεις απασχόλησης ε, από επιχειρήσεις οι οποίες επαναφέρουν θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα υπάρχει μικρότερη καθυστέρηση για τις επιχειρήσεις και αυτό θα δώσει τεράστιες ευκαιρίες ε, για την αύξηση της οικονομίας γενικότερα. Τα κράτη-μέλη μαζί με την Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα να βοηθήσουν την κεφαλαιοποίηση των εταιριών. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν την έκθεσή μου γιατί είναι ένα βήμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος περισσότερο φιλόξενου που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο κυρία Μακιντάιρ, διότι νομίζω ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε εκατομμύρια νέους ανέργους σε πολλά κράτη-μέλη. Σε πολλά κράτη-μέλη μπορεί να είναι από 5 έως 10% αλλά σε άλλα κράτη-μέλη είναι και 15%. Να μην πω ότι φτάνουν και το 50% σε ορισμένε περιοχέ. Θέλουμε λοιπόν ε, επιχειρήσεις που να είναι καινοτόμε, που να είναι στραμμένες προς το μέλλον και να δημιουργούν θέσεις απασχόληση. Και θέλω να πω ε, και να ευχαριστώ προ την Επιτροπή και τον Επίτροπο Ταγιάννη που ξεκίνησαν ε, μια σχετική έρευνα στον τομέα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσει. Πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολλές οι διατάξεις που ε, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε χάσει 8% ανταγωνιστικότητα στα τελευταία χρόνια ε, και εν πολύ οφείλεται αυτός στην γραφειοκρατία και σε διατάξεις που έχουν απομακρύνει θέσεις απασχόλησης από την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε συσχετισμό μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς ε, που ε, θέλουν να είναι ε, αυτοαπασχολούμενοι και πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα και να γίνουν εργοδότες και να αρχίσουν να προσλαμβάνουν προσωπικό. και θα πρέπει να δείξουμε ότι ε, για ε, κάποιον που ε, είναι αυτοαπασχολούμενος και αναλαμβάνει τον κίνδυνο να προσλάβει έναν υπάλληλο, έναν εργαζόμενο θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για να μπορέσει να κάνει τα σωστά βήματα. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ούτως ώστε οι νομοθετικές μας πράξεις να εξασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας και να μην δημιουργούν προβλήματα ε, και αντιθέτως ε, καταργούν θέσεις εργασίας. Ε, θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να γίνει ένα τεστ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως υπάρχει στην Γερμανία παραδείγματος χάρη και πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει νομοθεσία που θα είναι στραμμένη προς το μέλλον, θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης διότι θέλουμε νέους ε, που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν περισσότερα, να τους δίνουμε κίνητρα για να προσφέρουν περισσότερα και να δούμε ποια είναι αυτά τα κίνητρα ε, τα οποία θα οδηγήσουν κάποιον στο να γίνει αυτοαπασχολούμενος και ποια είναι τα κίνητρα που θα κάνουν ένα αυτοαπασχολούμενο να γίνει εργοδότης και να προσλάβει εργαζομένους. Να μην έχουμε ένα σύστημα που θα τιμωρεί ε, τους, ε, αυτούς που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία. Το πρώτο βήμα πάντοτε σχετίζεται με μεγάλους κινδύνους. Να μην το επιβαρύνουμε και με τιμωρία για αυτή την αποτυχία. Ας πάρουμε κάποιες ιδέες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το τομέα. Βλέπουμε ότι επιχειρήσεις, ιδίως στη χημική βιομηχανία, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με το REACH. Και έχει γίνει μια μελέτη που έχει δείξει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τηρήσουν ε, τις προδιαγραφές για να έχουν τις εγκρίσεις που απαιτούνται, δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό διότι θα απαιτούσε μεγαλύτερη οικονομική δύναμη για να ε, ανταποκριθούν. Έχουν επίσης ε, μεγάλα προβλήματα με τις επιστροφές ΦΠΑ οι επιχειρήσεις. Ε, καθυστερεί πάρα πολύ, καθυστερούν οι επιστροφές του ΦΠΑ. Θα χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα clearing που θα διεκπεραιώνει αυτά τα ζητήματα πολύ πιο γρήγορα, ούτως ώστε να μην είναι ε, δύσκολη η πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, όσον αφορά την βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Επίσης, να ληφθεί υπόψη και μια προσπάθεια μείωσης του διαστήματος πληρωμών σε διάφορους τομείς, στον κατασκευαστικό τομέα και σε άλλους τομείς για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν ιδέες που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούμπιχ αλλά πριν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Επιτροπό, υπάρχει μία ερώτηση μπλε κάρτα από την κυρία Τικάου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Τικάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ρούμπιχ το εξής. Το 2009 ένα πρόγραμμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου υιοθετήθηκε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μας πείτε αν λάβατε υπόψη αυτό το πρόγραμμα και πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσω του προγράμματος αυτού. Ευχαριστώ. Please, time for the answer. Απαντήστε. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Αυτό νομίζω ότι βρίσκεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που χρειάζονται κάποιες εγγυήσεις για επιχειρηματικό κεφάλαιο και γνωρίζουμε ότι ε, ε, με αυτό το μέσο μπορούμε να βοηθήσουμε τις, ε, τις επιχειρήσεις ε, και με ε, κάποια μικρή χρηματοδότηση να παράγουμε 25 και 30 φορές αποτελέσματα να παράγουμε αποτελέσματα 25 και 30 φορές μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο το οποίο επενδύουμε. Και νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να έχει περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο ε, Ταγιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τις, τους ε, κύριους ε, Ρούμπιχ και Μακιντάρ που μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε αυτή τη θητεία συζητώντας το θέμα της πραγματικής οικονομίας και προβλήματα που αφορούν 23 εκατομμύρια μικρές και μισές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η συζήτηση αυτή γίνεται στο τέλος μιας σκληρής δουλειάς ε, που έκανε η Κομισιόν μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν τέλει κατορθώσαμε να πείσουμε και το Συμβούλιο ότι είναι σημαντικό να δώσουμε στην Ευρώπη μια βιομηχανική πολιτική έτσι όπως ε, συνέβη στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου. Οι μικρές και μισές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα. Υπάρχει βέβαια και μεγάλη βιομηχανία, αλλά χωρίς ε, τις μικρές ε, και μισές επιχειρήσεις, όπως είπε και ο κ. Ρούμπιχ, δεν μπορούν να δημιουργηθούν αίσθηση εργασία και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την απασχόληση σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε κατά την απόψή μου. Ένα από τα μεγάλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να επιτρέψουμε στις σημερινές ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, την πρόσβαση αυτή. Το 23% ε, βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος και το 13% εργάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε το διοικητικό άχθος προκειμένου να άρουμε όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εργαστούν. Το έγγραφο για τη, που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν για την αναγέννηση της βιομηχανίας μιλά για τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η Κομισιόν θα έχουμε τρεις μέρες ε, ε, για να μπορεί να σχηματιστεί μία μικρή ε, και μεσαία επιχείρηση. Θα μειωθούν όλες οι προθεσμίες και η Κομισιόν εργάζεται και στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT για να εντοπίσει όλα τα κενά και τα αναποτελεσματικά μέτρα. Τον Ιούνιο η Κομισιόν θα παρουσιάσει μία ανακοίνωση για την κατάσταση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας REFIT και θα υπάρξει μία δημόσια διαβούλευση για να ξεκινήσει ένας περαιτέρω προβληματισμός για το θέμα προκειμένου στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT ε, να υπάρξει ένας πίνακας αποτελεσμάτων και να μπορέσει η Κομισιόν να προβεί σε μείωση του άχθους μέσω της νομοθετικής διαδικασίας και της εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ρούμπιχ ε, στην παρέμβασή του μας υπενθύμησε το top 10, ε, τα διοικητικά άχθη που εντοπίστηκαν μέσω Τη διαβούλευση. Προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσει και σε ό,τι αφορά το REACH, που είναι το πρώτο στον κατάλογο. Έχουμε μειώσει το άκρο τη καταχώρηση για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις από 35 μέχρι 90% διορίσαμε έναν πρέσβη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε παρουσιάσει προτάσεις απλούστευσης για έξι νομοθετήματα για την προστασία των δεδομένων, ασφάλεια των προϊόντων, δημόσιοι διαγωνισμοί κτλ. Και εργαζόμαστε για να δημιουργηθεί μια νέα θηρίδα για να διευκολύνουμε τις διαδικασίες σχετικά με το ΦΠΑ για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Επίσης, καλέσαμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν συστηματικά την αρχή του Think Small First σε όλες τις νομοθετικές πρακτικές τους. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προκειμένου να λειτουργεί το δίκτυο, όλα τα κράτη-μέλη έχουν διορίσει ένα πρεσβευτή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της εφαρμογής του Small Business Act και φυσικά όλο αυτό γίνεται υπό την ε, καθοδήγηση του δικού μου Γενικού Διευθυντή. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ε, απευθύνω άκληση στα κράτη-μέλη για να υπάρχει μια συνάφεια. Δηλαδή κάποια κράτη-μέλη όταν ε, καλούνται να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οπισθοδρομούν. Έχω κατά νου μια πρόταση που θα συζητήσουμε αύριο για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων σε άλλο κράτος μέλος. Καλό τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, να ε, σέβονται το γεγονότα. Τώρα ένα άλλο θέμα για την πρόσβαση στην πίστοση. Όπως ξέρετε στον κοινωτικό προπολογισμό έχουμε 150 δις για τη βιομηχανική πολιτική για πρώτη φορά 100 από τις περιφερειακά ταμεία 40 από τον ορίζοντα 2020 για την έρευνα και καινοτομία και 2,5 δισεκατομμύρια από το κόσμο το οποίο είναι το πακέτο που στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και Φυσικά υπήρξε τα τελευταία χρόνια πολύ στενή συνεργασία σε αυτά τα θέματα μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω και απόψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστήριξε τις προτάσεις της Κομισιόν καθώς προ προς την ίδια κατεύθυνση. Ο κύριος Ρούμπικ υπενθύμησε στην ομιλία του το θέμα των ελευθερών επαγγελματιών. Ε, τις προαλές υιοθετήσαμε ένα σχέδιο για τους ελευθερούς επαγγελματίες, ε, τους οποίους η Κομισιόν θεωρεί πραγματικούς επιχειρηματίες. Όπως ξέρετε, το έγγραφο που αναφέρεται στο επιχειρηματικό πνεύμα για πρώτη φορά προσδιορίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες ως επιχειρηματίες. Το σχέδιο δράσης προβλέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε κοινοτικό διαγωνισμό και να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική καινοτομία που οδεύει προ την κατεύθυνση του ποιου παράγει και δημιουργεί θέσει εργασία. Ξέρετε ότι έχουμε και το θέμα της εφαρμογής ε, της οδηγίας ε, για την καθυστέρηση των πληρωμών. Θα έπρεπε να είμαι αυστηρός και με τη δική μου χώρα, αλλά δεν πιστεύω ότι οι πολίτες δεν μπορούν ε, να μην βλέπουν ένα καλό παράδειγμα. Θα πρέπει οι πολίτε να πληρώνουν του φόρου, αλλά και τα κράτη θα πρέπει να πληρώνουν εντό προθεσμίας του προμηθευτέ του. Ένα άλλο έργο που ολοκληρώσαμε θετικά ήταν η Βασιλεία 3. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που εισήγαγε τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει στο Porting Factor που θα επιτρέψει χρηματοδότηση ω 1,5 εκατομμύριο ευρώ στι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει με πιο εύκολο τρόπο. Υπήρχε και το θέμα τη πρόσβαση στι διεθνεί αγορέ. Ε, και αυτό νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βγουν στις διεθνείς αγορές. Ε, υπενθυμίσω ότι μόνο το 13% μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος ε, για την ε, δυναμική και την ποιότητα των όσων παράγουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ο επόμενος μάλλον, είναι η κυρία Ντρέσ Μπαρέα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Λοιπόν, ας περάσουμε στην ε, κυρία Κάντερμπαχ από την Επιτροπή Ρέτζη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συνεχίζω αμέσω μετά την παρέμβαση του Επιτρόπου και χαίρομαι ε, που ακούω ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε δανεισμό και σε χρηματοδοτικά όργανα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και από την πλευρά των περιφερειών να πούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιχειρηματικό πνεύμα, ε, να τους δίνουμε κάθε δυνατότητα που είναι δυνατόν να τους προσφέρουμε. Υπάρχει, ε, υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνουν πολλές ε, δυνατότητες, καλύτερη ενημέρωση ε, για δικτύωση, για δημιουργία της επιχείρησης, για πρόσβαση σε νέες αγορές όπως είπατε και σημαντικό για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι να τις βοηθήσουμε και τα πρώτα πέντε χρόνια γιατί αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της ανεργίας, να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης στους νέους και αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ε, βοηθούν άλλους νέους ε, να βγουν στην αγορά εργασίας. Είναι μια δυνατότητα που πρέπει να προσφέρουμε στην νεολαία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, η κυρία Σάγια για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, στο ΕΛΚ, η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερως, γιατί πρόκειται για την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό συνδέεται άμεσα με την φορολογία και ε, προάγει και την ευημερία. Έχουμε εξετάσει το πλαίσιο και προγράμματα όπως ε, το Small Business Act και επιχειρηματικότητα 2020. Τώρα, αν το εξετάσουμε σε εθνικό επίπεδο, βλέπουμε ότι δεν διατίθονται όλοι, όλες οι δυνατότητες ε, για τις μικροπιστές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο. Δεν έχουν δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις ε, το δικαίωμα να κάνουν τέτοιου είδους αιτήματα. Έχουμε το πρόγραμμα Refit, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τώρα όμως πολύ συγκεκριμένα, η σύσταση μιας ε, επιχείρησης θα έπρεπε να καταστεί πολύ πιο εύκολη και απλή και εκεί θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την αρχή της ενιαίας θηρίδας. Αυτή τη στιγμή διερχόμεθα μια οικονομική κρίση Παρά το γεγονός ότι έχουμε ε, διάφορα ε, χρηματοοικονομικά μέσα στη διάθεσή μας και πάλι όμως ε, αυτός ο κλάδος είναι από τους πιο σημαντικούς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Ντεμπάκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την οικονομία μας. Συζητώντας με τον επιχειρηματικό κόσμο, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα μπορούν να επανέλθουν και τα οποία κάποια μπορούμε να τα αποδεχθούμε, κάποια πρέπει να τα στείλουμε πάλι πίσω και κάποια πρέπει να τα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Το πιο σημαντικό ε, είναι η κατάλληλη κατάρτιση. Απαιτείται λοιπόν η κατάρτιση και για τα άτομα τα οποία θα απασχοληθούν σε αυτέ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ σημαντική ενεργεία των νέων στην Ευρώπη, όμω βλέπουμε ότι σε πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει υπάρχουν διαθέσιμες θέσει εργασία, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση αναγκών και ζήτηση. Το δεύτερο τμήμα, σημείο που θα θέλαμε να θίξουμε θα ήταν η νομοθεσία που έχουμε εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιε φορέ πρέπει να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη νομοθεσία μα για τι μικρέ, μεσαίε ή μεγάλε επιχειρήσει. Και εδώ νομίζουμε ότι έχει, έχουν αναπτυχθεί καλέ προτεραιότητε ε, για την ε, κάλυψη κάποιων κενών και το τελευταίο τμήμα βεβαίως αφορά την χρηματοδότηση. Αν θέλουμε αυτές οι επιχειρήσεις και θέλουν αυτές οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, χρειάζονται χρηματοδότηση όχι μόνο μέσω ε, τραπεζών αλλά και μέσω αγορών Και θα πρέπει να επιστρέψουν προσοχή σε αυτό το γεγονό, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε άλλες μορφές χρηματοδότησης αυτές οι επιχειρήσεις και έτσι να βελτιώσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κριστίνα Μόρβαη. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα. 24 βουλευτές Συγχαρητήρια. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα γιατί εδώ μιλάμε για μικρομεσαίε επιχειρήσει, μιλάμε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ελπίζω στην Ουγγαρία κάποια μέρα οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι τη λήψη αποφάσεων να κατανοήσουν ότι δεν πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα. Η δημιουργία θέσεων απασχόληση αυτό το θέμα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι Ούγγροι εργαζόμενοι να εργάζονται για πολυεθνικές, χωρίς δικαιώματα και με ε, πολύ χαμηλό μισθό. Η δημιουργία θέσεων απασχόληση σημαίνει ότι δίνουμε νέες ευκαιρίες σε νέους να ε, βρουν μια πραγματική θέση εργασίας και πρέπει να δούμε τι ακόμα πρέπει, να γίνει για να γίνουν οι Ούγγροι πραγματικοί πολίτες αυτού του κόσμου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το σημείο 54 του κειμένου που μιλά για τη δυνατότητα που έχουν, ε, για τις δυνατότητες που έχουν επιχειρηματίες και ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με, τη δυνα... με τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Θα πρέπει να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε όσους τα χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Θα ξεπεράσουμε τώρα στη διαδικασία Κατσδιάη και θα δώσω το λόγο στην κυρία Παναγιώτοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μακιντάρ για την εκθεσή της. Μας περιγράφει την κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αν ε, θέλουμε να έχουμε αναπτύξει στην Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ε, υπάρχουν διάφορες διοικητικές και οικονομικές δυσκολίες ε, και μόνο 17% των στην Ευρώπη πιστεύουν ότι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις στη διάθεσή τους. Ε, υπάρχει το θέμα του χρόνου και γι' αυτό η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, στην εμπειρογνωμοσύνη και σε διάφορες μορφές επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι για τους επιχειρηματίες. Θα πρότεινε το 2017 να διακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Επιχειρηματικότητας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και ελπίζω ότι αύριο μετά την ψηφοφορία αυτή η πρόταση θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόμασιτς. Είμαι από την Κροατία όπου το επιχειρηματικό πνεύμα έχει υποφέρει από αστάθεια και λόγω της ε, μη προβλεψιμότητας κυβερνητικής πολιτικής υποστηρίζω τα όσα υπόθηκαν. Ενώ ακούγαμε πολιτικές υποσχέσεις για ανάκαμψη και ανάπτυξη, ε, ουσιαστικά είδαμε το αντίθετο αποτέλεσμα και τέτοιες εκθέσεις μου δίνουν ε, την δυνατότητα να είμαι αισιόδοξη γιατί το μόνο που έχουμε δει είναι ε, υπερβολική και νομοθεσία και φόροι, ε, πράγμα που έχει επίπτωση στην νοοτροπία στη χώρα μου. Κάθε πολιτικό πείραμα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στη χώρα μου. Υπάρχουν Πολλέ χιλιάδες άνεργοι και περαιτέρω γραφειοκρατία. Πού θα πάει αυτό, ο κύριος Μπενιόν. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σημερινό οικονομικό κλίμα ζητά να δούμε πολύ προσεκτικά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και ανάπτυξη. Η έκθεση αυτή συνεισφέρει σημαντικά σε αυτή τη συζήτηση, καθώς επικεντρώνεται στη σημασία τη επιχειρηματικότητα Κάτι που και εγώ έχω κηρύξει ότι θα πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια και επίση πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα για τι επιχειρήσει. Κυρίω ε, πρέπει να εξετάσουμε το διοικητικό άχθο επί των επιχειρήσεων. Ε, Όμω ε, από τα αριστερά προσπάθησαν κάποιοι να αφαιρέσουν πολλά σημαντικά στοιχεία από την έκθεση. Οι πράσινοι φαίνεται να μην πιστεύουν ότι πρέπει να δυσφαλίσουμε τα συστήματα εκπαίδευση. Πρέπει να απαντάνε στι επιχειρηματικέ ανάγκε μέσω των, δεξιών, των, των δεξιοτήτων STEM και οι σοσιαλιστέ φαίνεται να πιστεύουν ότι οι συμφωνίε των κοινωνικών εταίρων πρέπει να υποκείται σε δημοκρατικό έλεγχο. Θα πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική ένωση που να έχει στο επίκεντρο το θεματολόγιο τη καλύτερη νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εδώ όλα τα στοιχεία αυτή τη έκθεση κατά νου. Ευχαριστώ κύριο Ράνσοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Ταγιάννη, το εξή. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια χρηματοδοτικά μέσα θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για να γεφυρώσετε το χάσμα που υπάρχει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν πάνω από 70% των θέσεων απασχόλησης αφενός, από την άλλη πλευρά έχουν μόνο 4% μερίδιο στην έρευνα και ανάπτυξη. Εδώ υπάρχει ένα χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί. Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να αρθεί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν και σωστό τεχνολογικό εξοπλισμό. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρία Νικόλ Σινκλέρ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Μακιντάρ για τις προσπάθειές της για την έκθεση αυτή. Και όπως και εκείνη και εγώ επιθυμώ το καλύτερο δυνατόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την ικανότητά τους να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Το 43% των απασχολουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι η κυρία Μάκιντάρ πιστεύει ότι αυτό μπορεί να το επιτύχει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβούμαι ότι δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Μαζί με τον κύριο Φιλ Μπάνιον, το 2009 στο Μπέρμιγχαμ, είδαμε την Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων που είπαν στο μανιφέστο τους ότι δεν θέλουν άλλη νομοθεσία που να έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν άλλη γραφειοκρατία. Κυρία Μακιντάιρ, θα έπρεπε να φροντίσετε να μειώνετε τη γραφειοκρατία και ο κύριος Ρούμπιχ που έλαβε το λόγο δεν έχει φροντίσει να μην χάνουμε θέσεις απασχόλησης για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τον κύριο Ταγιάννη να κλείσει τη συζήτηση αυτή τώρα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει γενική συνένεση για τη σημασία που πρέπει να δώσουμε τα επόμενα χρόνια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να καταπολεμήσουμε την κρίση και να δώσουμε προοπτική εργασία στους νέους. Θέλω να σταθώ στο θέμα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και στην πρόσβαση στην πίστοση. Εμείς αποφασίσαμε 150 δισεκατομμυρία να τα διοχετεύσουμε στην πολιτική της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και αυτά θα προέρθουν από τα περιφερειακά ταμεία το 40% τα 40 από τον ορίζοντα 2020, 2,5 δις από το κόσμο. Μπορώ να σας πω, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διοχετεύσει το, 25, το 20% συγγνώμη στις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Κατόπιν ε, δώσαμε μία μάχη για το κόσμο, για τη διεθνοποίηση, για τον κλάδο του τουρισμού και για το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, μόνο για τις μικρομεσαίες. Επίσης υπάρχει μεγάλη δέσμη που είχε προτείνει η Κομισιόν μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μπλοκαριζόταν από το Συμβούλιο γιατί πολλές φορές ε, γίνεται προσπάθεια να αποκρυπτούν οι πραγματικές ευθύνες ε, κάποιων κρατών μελών. Ε, κάποιοι διαμαρτύρονται ότι υπάρχει υπερβολική κοινοτική γραφειοκρατία και κατόπιν όταν εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε αυτή τη γραφειοκρατία, οι συγκεκριμένες χώρες αντίθετα υπερασπίζουν την γραφειοκρατία και το γραφειοκρατικό άχθος. Δυστυχώς ε, η δέσμη μέτρων έχει μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ασκούμε μία πίεση, γιατί αν θέλουμε να καταστήσουμε πραγματική την πρόταση αυτή της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενθύσεων ε, που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση για μια ακόμη φορά μα έδειξε πόση συμφωνία υπάρχει μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου για την προστασία του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα βγούμε από την κρίση μόνο αν μιλάμε για τη μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά θα βγούμε από την κρίση μόνο αν είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία να αναπτύξουμε την αγορά. και να ακολουθήσουμε την ε, θεμελιώδη γραμμή, ε, να δημιουργήσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η αγορά είναι ένα εργαλείο για να έχουμε κοινωνική πολιτική και αυτό το κάνουμε αν συνεχίζουμε να βοηθάμε την βιομηχανική πολιτική και να προωθούμε την πολιτική υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία και θα αποτρέψουμε περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο τη κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, κύριε Μακιντάιερ. Έχετε το λόγο. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ βασικά στοιχεία σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις, ιδίω οι μικρομεσαίες, θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη, γνώσει και τεχνογνωσία, να έχουν πρόσβαση ε, σε χρηματοδότηση μέσω ενιαστηρίδα ε, και ε, διαδικτυακών πυλών. Δεύτερον είναι σημαντική η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος από μικρή ηλικία και στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Και κύριε Ρούμπρεκ, χαίρομαι ιδιαίτερως που θίξετε αυτό το ζήτημα για το πώς πρέπει πραγματικά να διδάξουμε τους, τους νέους μας ε, για την επιχειρηματικότητα. Να συγχαρώ και στους αδέλφους που είπαν, ε, ε, έκανα την πρόταση να υπάρξει η έτος επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και για τον κύριο Τομάτσικ να μειωθεί η γραφειοκρατία για να αφήσουμε τις κροατικές επιχειρήσεις να διαπρέψουν. Είναι πολύ σημαντικό. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει μας λένε ότι η ευρωπαϊκή αγορά με τα 500 εκατομμύρια πελάτες και καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ελκυστική ε, για τις μικρές επιχειρήσεις και εμεί, ω νομοθέτε, θα πρέπει να μειώσουμε την γραφειοκρατία και το άχθο που επομίζονται οι επιχειρήσεις. Αν είστε ένα επιχειρηματία που έχει μια μικρή επιχείρηση, κάνετε όλη μέρα δουλεύετε τόσο σκληρά, ε, κάνετε την πραγματική δουλειά και μετά πρέπει να δείτε το λογιστή, το δικηγόρο και το καθεξή, να του δείτε όλου αυτού το βράδυ. Δουλειά μα είναι να τα κόψουμε όλα αυτά, ούτω ώστε ο επιχειρηματία να μπορεί να επικεντρώνεται ε, στη δουλειά του, που είναι η δημιουργία πλούτου, η ανάπτυξη και ε, το πώ θα μπορέσει να δώσει δουλειά σε περισσότερου εργαζομένου. Επομένω, Στηρίζω την έκθεσή μου και ελπίζω όλοι να ενωθούμε για την ε, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, την αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για να επιτρέψουμε την επιτυχία ε, των επιχειρησιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτού του θέματος για την έκθεση McIntyre. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο για αυτή την έκθεση. Α, συγγνώμη. Αύριο στις 6 το απόγευμα, λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να ρωτήσω σε πόσους δεν δώσατε το λόγο που τον ζήτησαν στη διαδικασία Catch the Eye. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ σήμερα ξύπνησα 5.30 ώρα το πρωί, είναι 10 η ώρα το βράδυ, θα έπρεπε να μας δώσετε δυνατότητα να μιλήσουμε. Γιατί τις περισσότερες φορές παραπονιέστε ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέλη ε, στην Ολομέλεια. Αλλά βέβαια δεν είναι δίκαιο να μην τους δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πόσοι ε, ζήτησαν το λόγο και δεν του το δώσατε. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο αριθμό, καταλαβαίνω. Όπω θα θυμάστε, λέει ο Πρόεδρο, κύριε Κέλλη, οι κανόνε ότι ε, κατά μέγιστο βαθμό πέντε ομιλητέ μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Έδωσα το λόγο σε πέντε από του εννέα. Συγγνώμη, αλλά δεν ήσασταν ο πρώτο από το ΕΛΚ που ζήτησε το λόγο. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Η παρεμβάση του ενό λεπτού. Η κυρία Έντιτ Μπάουερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μαλίνα Εντβίγκ, ε, φοιτήτρια από την Ουγγαρία, ε, διώκεται εδώ και 7 έτη.